Έχουμε τις της ψήφου και θα πρέπει όλοι όσοι το επιθυμούν να μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Ξεκινάμε τις, με τις ε, για την έκταση πυρή. Ο συνάδελφος Αστροβίτσιος έχει το λόγο. Mr. Chairman. Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της εκθέσεως και ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ήδη έχει εγκριθεί ένα ψήφισμα για την Τουρκία σε σχέση με το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Σε εκείνο το ψήφισμα τονίζουμε ότι η Τουρκία παραμένει στη δικοστήρα της Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είπαμε ότι προβληματιζόμαστε βαθιά όσον αφορά με πάρα πολλές ασυμβατότητες όσον αφορά την προσχώρηση για τα σχετικά προγράμματα και είπαμε ότι θέλουμε προσωρινό πάγωμα των σχέσεων. Αλλά από τότε η κατάσταση επιδεινώθηκε και ε, συνεχίζει να υπάρχει μονοκρατορία στην χώρα. Έχουμε ε, συλλήψεις, ε, δημοψήφισμα για αντισυνταγματικές ε, μεταβολές στο πολίτευμα και επίσης έχουμε και φήμωμα των ΜΜΕ. Άρα δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτή την κατάσταση. Εάν η δέσμη συνταγματικών μέτρων εφαρμοστεί όπως έχει τώρα, θα πρέπει να διακόψουμε τις συνομιλίες προσχώρησης με την ε, χώρα. Όπως επίσης να σταματήσει και η προενταξιακή χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφος Άνων ναι, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ των υστέρων η προσέγγιση ε, φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο σωστή. Από την αρχή είχαμε πει ότι ε, το να γίνει μέλος δεν είναι στο θεματολογείο μας, έχουμε έναν άλλο τρόπο, αλλά τελικά αυτό το οποίο έγινε είναι ότι δώσαμε μια υπόσχεση που δεν είχαμε ποτέ την πρόθεση να την τηρήσουμε. Οπότε, ε, επομένως, ε, επικράτηση, απογοήτευση ε, όλα αυτά τα οποία έγιναν στη χώρα της Εξελίξης δεν λέω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ίσως δεν είναι ούτε τώρα σωστό εάν τώρα θέλουμε να προσπαθούμε να βρούμε μια βιώσιμη συμφωνία. Αναγνωρίζουμε ότι αξίζει μια ελεύθερη αγορά με την Τουρκία. Είναι στρατηγική δοτικό εταίρος η Τουρκία, αλλά δεν μπορεί να έχουμε κάποιο άλλη πολιτική ολοκλήρωση. Είναι σημαντική χώρα, μεγάλη χώρα. Οπότε αν τα καταφέρουμε, τότε μπορεί να γίνει παράδειγμα προσμίμηση στις γειτονικέ χώρες. Ευχαριστούμε κύριο Νταμπαύσκη. Έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαρητήρια στην κυρία Πύρη, τη συνάδελφό μας, για την εξαίρετη έκθεσή της. Αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η έκθεση αυτή, γιατί αντεκατοπτρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, εγώ καταψήφισα γιατί η έκθεση δεν μιλάει για την ε, αλλαγή της ε, κοσμικής ε, Τουρκίας του Κεμάλ σε ε, θρησκευόμενο κράτος. Πρόκειται για μια στροφή στο Ισλάμ της χώρας και η Τουρκία βλέπουμε ότι αναμειγνύεται στις υποθέσεις ε, πολλών χωρών στην περιοχή, της Βουλγαρίας, της χώρας μου για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι καλό. Οι σχέσεις με την Τουρκία πρέπει όντως να παγώσουν. Δεν μπορεί να είναι σύμμαχός μας. Είναι μια Ισλαμική δικτατορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σαμπόσκα τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, συμφωνώ με τις δύο τροπολογίες του ΙΕΝΕΦ. Η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και εδώ έχουμε να κάνουμε και με την συνεννόηση, την καλή συνεννόηση καθολικών και μουσουλμάνων. Η Αγία Σοφία πρέπει να παραμείνει μουσείο. Δεν υπερψήφισα όμως τις τροπολογίες αυτές γιατί είναι σχετική κατάσταση στην Τουρκία. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία είναι καθοριστικά για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση το κείμενο αυτό πρέπει να υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Τουρκίας τις υποχρεώσεις της και να τη θυμίσει επίσης και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. Όταν θα δείξει καλή θέληση τότε θα περάσουμε σε πιο καθόδη ζητήματα. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρσκα. Τελειώσαμε την έκθεση Πύρη, περνάμε την έκθεση Κούκαν. Και Καρταρούμπια. Ο κύριος Όστρεβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ αυτού του είδου του επενδυτικού σχεδίου πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το ότι είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να μείνει πηγή υποστήριξη για αυτέ τι χώρε. Χαίρομαι ότι οι ιδιωτικέ επενδύσει θα χρησιμοποιηθούν στην ε, Αφρική και επίσης ε, ανατολικά και νοτιώς των συνόρων μας σαν μέρος της στρατηγικής να συγκρατηθεί η μετανάστευση έτσι θα χτυπήσουν τη σύνδεση μετανάστευση, επασχόληση, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διευκόλυνση της ε, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Οπότε έχουμε τώρα το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη και επίσης ε, παρέχονται εγγυήσει ότι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρησιμοποιηθεί για να επενδύσει επενδύσει σε ιδιωτικό και δημοσίου τομέα και θα διαχειριστούμε και τον κίνδυνο. Οπότε τώρα θα ε, υπάρχουν αρκετέ ε, ε, επενδύσει με αυτό το μέσο το οποίο εγκρίναμε. Και έτσι θα υπάρξει βιώσιμη τεχνική αρρωγή σε όλε τι χώρε που την χρειάζονται. Και σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αγγιλέρα Γκαρτία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ Αυτή τη εκδοχής και να λέω το λόγο για αυτό το Ταμείο, το Ταμείο της Ευρώπη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί οπωσδήποτε έτσι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη φτώχεια τη αδικία και τη μετανάστευση. Έχουμε περίπου 44 εκατομμυρίων για τις επενδύσεις σε Αφρική και τις γειτονιάσουσες χώρες. Ε, επομένως έτσι θα αντιμετωπίσουμε το βασικό πρόβλημα που έχει η Αφρική για να αντιμετωπίσουμε και κάποιες αδικίες. Θέλω τώρα να τονίσω κάποια θετικά σημεία που είναι πολύ σημαντικά για το Ταμείο. Η μνήμα για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, την ανθεκτικότητα, την αξιοπρεπή απασχόληση και κρίζωση της ε, φτώχειας. Ότι θα πρέπει να καλυφθεί η Συμφωνία των Παρισιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι στόχος αυτού του ταμείου και επίσης να έχουμε και αυτή την ιδιαίτερη διαφύλαξη για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. Τέλος, το ότι στο κείμενο αναφέρεται και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, επιτυχίες για το Ταμείο. Σας ευχαριστώ, κύριε Αγγιλέρα Γκαρσία και περνάμε λοιπόν τώρα Ολοκληρώθηκαν έτσι οι αιτιολογίε ψήφου για την έκθεση Κούκαν και να περάσουμε τώρα στι αιτιολογίε ψήφου για την έκθεση του κ. Άντερσον. Η κυρία Σόντροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίναμε την νομοθεσία αυτή σήμερα Πρόκειται για την ενσωμάτωση της ηθίκης του Μάρακες που προβλέπει την χρήση προστατευόμενων έργων και άλλων προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών κλπ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί έτσι και τα άτομα αυτά μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή. Φυσικά χρειάζεται συνεργασία των χωρών μελών Χρειάζονται και εναλλακτικέ μέθοδοι επίσης, στο Μπράιλ, σε, πιο, σε διαφορετική διάσταση. Πάνω από 20% των έργων υπάρχουν ήδη διαθέσιμα, αλλά μένει το 80%. Αν το πετύχουμε και αυτό, έτσι θα έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες τα άτομα αυτά να έχουν εκπαίδευση και το εμπόριο επίσης θα ενισχυθεί. Αλλιώ τα άτομα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθόλου τα προστατευόμενα έργα. Πιστεύω ότι όταν έρθουν αυτά τα εμπόδια θα διευκολυνθεί πάρα πολύ η ζωή τους. Ευχαριστούμε κυρία Σόντροβα. Στέλλερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και χαίρομαι που σήμερα είμαστε πιο κοντά στην κύρωση της συνθήκη του Μαρακές. Η δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διευκόλυνση στην πρόσβαση των τυφλών σε τέτοια αγαθά είναι ένας αγώνας που έχουμε δώσει εδώ και καιρό και επιτέλους τα καταφέρνουμε. Είναι ένα από τα θετικά στοιχεία είναι η αποζημίωση, διότι πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 21 τη σύμβαση του ΟΙΕ για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά δεν υπάρχει και καμία απόδειξη ότι χρειάζεται αντιστάθμιση γιατί υπάρχει κάποια απώλεια από τις επιχειρήσεις και ούτε φαίνεται αλλάζοντας το μορφότυπο να υπάρξει ζημιά στους εκδότες. Πρέπει να μπορούν λοιπόν όλοι να έχουν πρόσβαση και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε με την κύρωση της σύμβασης αυτής του Μαρακές. Πάντως ελπίζω οι χώρες μέλη να κυρώσουν ώστε να προχωρήσει η σύμβαση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Στήλερ. Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι τελικέ ψήφου για την έκθεση του κυρίου Άντερσον και τώρα να ακούσουμε τη συντηλογή τη ε, ψήφου για την έκθεση δένση. κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι βήμα προ την εμπρό όσον αφορά μια βιώσιμη ανάπτυξη για την Ευρώπη. Οπότε γι' αυτό και ψηφίσαμε υπέρ όλα αυτά. Να τονίσουμε ότι θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξο το κείμενο και να έχουμε δεσμευτικού στόχου πρώτα-πρώτα για την εξοικονόμηση ενέργεια για να μπορέσουμε να έχουμε ε, κάποιο είδους ε, αλλαγή στο βιομηχανικό περιβάλλον των ε, πόλεων, να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος, γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για τις διάφορες ρηπαντικές ουσίες που αφορούν το νερό και το έδαφος. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο η ανακύκλωση. Εμείς προτείναμε κάποιες τροπολογίες που δεν πέρασαν όσον αφορά τα απορρίμματα. Ε, να αναβαθμιστεί ε, η χρήση του, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό να καλυφθεί από το ΕΦΣΙ. Με αυτή την πρόταση γίνεται ένα άλμα προς τα εμπρός. Νομίζω διαλέξαμε την σωστή λύση. Σας ευχαριστώ. Στην αδερφή μάτω, η κυρία Αγγιουλέρα Γκαρσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για σημαντική έκθεση στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω να σα πω στην επεξήγηση του ψήφου ότι προτιμώ το πώ τελικά κατέληξαν τα πράγματα στην Ολομέλεια ε, σε σχέση με τα όσα είπαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή δράση για την βιωσιμότητα της Κομισιόν. Και αρχικά αυτά τα οποία εγκρίθηκαν στην Επιτροπή ήταν πράγματα άδικα για την ε, γεωργία. Αυτά διορθώθηκαν και ψήφισα υπέρ και σας τονίζω ότι η κοινή αγροτική πολιτική με την τελευταία μεταρρύθμιση ε, υπέστη κάποιες αλλαγές, μια στροφή πράσινη υπέρ του περιβάλλοντος. Έγινε αυτό το πρασίνισμα, το greening και αυτό προϋποθέτει και τέλος να έχει συνέπεια σημαντικές προσπάθειες για τους ε, γεωργούς Άρα δεν είναι κατά του περιβάλλοντος η Ευρωπαϊκή Γεωργία και έχουμε και το θέμα της ανταγωνιστικότητας και του ανταγωνισμού μάλλον με τα προϊόντα των τρίτων χωρών που δεν σε αυτό το περιβάλλον όπως εμείς. Σας ευχαριστώ συνάδελφα Αγγιλέρα Γκαρσία και τώρα έχουμε τον συνάδελφο Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, Ακολούθησε την οδό τη αποχής για την έκθεση γιατί δεν λέει τίποτα και ο ε, ο όρος της βιωσιμότητας δημιουργείται, χρησιμοποιείται με τόσο ευρεία έννοια που δεν σημαίνει τίποτα τελικά. Η έκθεση αυτή λοιπόν αποτελεί τίποτα παραπάνω από μια ανταλλαγή απόψεων. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που αναφέρονται για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και σε ό,τι αφορά τις περιοχές της Υπέτρου. Ε, δεν έχουμε άλλα ζητήματα τα οποία επίσης αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Τα εργαλεία για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη δεν λειτουργούν. Και δεν νομίζω ότι η χρήση των ε, κονδυλίων ε, του φορολογούμενου τελικά οδηγεί σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Λοιπόν, θεωρώ καλές προτάσεις και γι' αυτό δεν υποστήριξα την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Τζεμπάσκη. Η, κυρία, η κυρία Γκραπίνη δεν είναι εδώ, γι' αυτό το λόγο έχει ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο ίδιος ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, πολλά μένουν ακόμα να γίνουμε για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο για μας και τις επόμενες γενιές. Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στη στρατηγική 2020 του ΟΗΕ που απαιτεί τη στήριξη όλων των χωρών μελών και της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε λοιπόν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για μια συζήτηση για τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και δημιουργεί και έτσι και ένα πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, άρα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή λοιπόν μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου μας που είναι ένας καλύτερος κόσμος στο μέλλον. Ευχαριστούμε ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Οι στόχοι βιωσιμότητας στο ΟΕ καλύπτουν όλες τις πτυχές. Οι στόχοι του 2030 μιλούν για βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030 για όλους. Και αυτό είναι ένας στόχος που πρέπει όλοι να συμμεριζόμαστε. Ανθρώπινη εξωπρέπεια, σταθερότητα, ένας υγιής πλανήτης, δικαιοσύνη στην ε, κοινωνία, αυτή είναι η στόχη του 2030, γι' αυτό και υπερψήφισα. Οι στόχοι αυτή βιώσιμης ανάπτυξης θα διασφαλίσουν ανάπτυξη και θα διασφαλίσουν και μελλοντικές ε, σωστές πολιτικές. Πρέπει να φροντίσουμε το 2030 να έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Επίσης, Θέλω να σας συγχαρώ, Πρόεδρε, για τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύσατε σήμερα, σε αντίθεση με αυτά που είπε κάποιος άλλος ομιλητής νωρίτερα. Εγώ πιστεύω ότι η ψηφοφορία αυτή διεξάχθη πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και mm-hmm. για τα, για τα καλά λόγια. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν για την έκθεση του συναδελφού Ντάτς. Να περάσουμε στην τελευταία έκθεση στην έκθεση Ομαντζή και τώρα έχουμε τον συνάδελφο Νέκοφ. Πρόεδρε, μιλούμε τώρα τι γίνεται με αυτές τις εξόχους από τις περιοχές της ε, Ένωσης, αλλά επίσης και τις ε, ορεινέ περιοχές αυτές είναι πώς το ζήτημα της Ένωσης. Έχουν κάποιες ε, ιδιομορφίες, οπότε και βέβαια έχουν πιο δύσκολη πρόσβαση στην αγορά. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερου κάθε καθεστώτος και μεταχείρισης και να αναδέχονται ευκολότερα την χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό. Η πολιτική συνοχή προσφέρει ευκαιρίες σε αυτές τις περιοχές και άρα θα πρέπει αυτά να ισχύουν και μετά το 2020. Αυτές οι από κεντρες ορεινές περιοχές ε, παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επομένως θα πρέπει να είναι απλοί οι κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τα προγράμματα ποιοτικής παραγωγής και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει ενημερωτική εκστρατεία και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτό αποτελεί ευκαιρίες για την ζωή των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Νέκοφ, και έτσι ολοκληρώθηκαν και οι επιλογέ τη ψήφου για την εκκλησία Μόζη. Και έτσι ολοκληρώσαμε και την ημερήσια διάταξη. Και θέλετε, η σύνοδος μέχρι τις 3 ε, η ώρα το απόγευμα. Καλό μεσημέρι.